παρθενική σας εμφάνιση εδώ. Έχει δίκιο ο Μπαρτστάς. Δεν σας ε, ε, καλωσόρισα όπως αρμόζει. Ε, μπράβο σας. Πάμε στην επόμενη μελέτη. Δημοκρατική λογοδοσία και έλεγχος του προϋπολογισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιροποίηση, ενημέρωση. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Δεν ξέρω ποιο είναι. Α, είναι η κυρία Άκερμαν. Έχει έρθει πανελειμμένα. Δεν έβλεπα το όνομά σας. Και προχωράει και η ηλικία μου και δεν βλέπω κιόλα τόσο μακριά. Okay, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, ανέφερε η Πρόεδρος, ε, πρόκειται για επικαιροποίηση προηγούμενης ε, έκθεσης. Δεν είναι δηλαδή μια έκθεση από την αρχή. Θα καλύψω σημεία που ενδεχομένως να έχουν καλυφθεί στο παρελθόν, γιατί εγώ ήρθα προς το τέλος των παρουσιάσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Άκουσα δηλαδή πολύ παρόμοια ζητήματα ορισμός των ΜΚΑΟ μικρών, ποιοι είναι οι κύριοι δικαιούχοι, αποδέκτε δηλαδή ευρωαϊκών κονδυλίων, διαφάνεια του Μητρώου και η παρακολούθηση των βασικών συστάσεων της προηγούμενης μελέτης. Προτού προχωρήσω, νομίζω ότι η βασική εστίαση της ενημέρωσης αυτής, της επικαιροποίησης αυτής, ήταν ότι η ποιότητα και η προσβασιμότητα στα δεδομένα χορηγίας από ευρωπαϊκά κονδύλια βελτιώνεται, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Η πρώτη φορά που το είδαμε, το εξετάσαμε το θέμα αυτό ήταν το 2010 και ξανά το 16-17 Θυμάμαι ότι το 2010 ήταν αδύνατον να καταλάβει κανείς από πού προέρχονταν τα διάφορα δεδομένα, διάφορες γενικές διευθύνσεις κομισιών και δεν ήταν καν σαφές αν αναφερόμασταν στις ίδιες ΜΚΟ, άλλο τμήμα τους, άλλη οντότητα υπό την ίδια οργάνωση, υπήρχαν διάφορες ασυνέπειες ονοματολογίας. Εκεί πραγματικά είδαμε σημαντικές βελτιώσεις. Τώρα, για το σημείο αυτό, ορισμός των μη κάπα ομικρων Υπό τη δική μας οπτική. Δεν σημειώσαμε κάποιες εξελίξεις από την προηγούμενη μελέτη. Και στην οποία είχαμε σημειώσει ότι ένα βήμα προς τα εμπρός θα ήταν να παρακάμψει κανείς την ταξινόμηση των ΜΚΟ και να συμφωνήσει τουλάχιστον σε κατηγορίες τέτοιων οργανώσεων μεταξύ τουλάχιστον των διευθύνσεων της Κομισιόν. Διότι οι διάφορες υπηρεσίες των, της Κομισιόν χρησιμοποιούν, συνεργάζονται με διαφορετικές κατηγορίες και ακόμα αν την ταξινομήσουμε ως ΜΚΟ θα έπρεπε να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ του πώς τις κατηγοριοποιούν οι διαφορετικές υπηρεσίες της Κομισιόν. Προκειμένου κανείς να μπορέσει να προβεί σε μια ορθή πολιτική ανάλυση. Υπάρχει όμως ασυμβατότητα μεταξύ τραπεζών δεδομένων της Κομισιόν. Η τράπεζα δεδομένων LIFE είχαμε σημειώσει και από προηγούμενη μελέτη που ήταν μια συνοπτική, μια μεγάλης κλίμακας τράπεζα δεδομένων που συμπεριελάμβανε 16 κατηγορίες οργανώσεων και ιδρύματα και ιδρυμάτων οι οποίες τελικώς συμπιέστηκαν στο σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας σε δύο κατηγορίες, είτε κερδοσκοπικές, είτε μη κερδοσκοπικές ή δεν έγινε κάποια άλλη προσπάθεια ανάλυσης κατηγοριοποίησής τους κάποιες κατηγοριοποιούνται από μόνες τους και σε σχέση με πανεστημιακούς φορείς, ε, δηλαδή ακόμα και τμήματα ακαδημαϊκών φορέων μπορεί να αυτονομάζονται μικά και σε κάποιες χώρες από ό,τι κατάλαβα δεν είναι καν δυνατόν ένας ακαδημαϊκός φορέας, ένα πανεστημίο να κατηγοριοποιηθεί, να καταχωριστεί ως μη Επομένως, σε απάντηση του τι είναι μη επειδή των ορισμών των κρατών μελών ακόμα έχουμε ένα περίπλοκο σύνολο όπου κάποια ακαδημαϊκοί φορείς συμπεριλαμβάνονται σε κράτη-μέλη, άλλοι όχι, σε άλλα κτλ. Ή, ακούσαμε ότι Κομισιόν ε, λαμβάνει υπόψη της μόνο τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, αλλά κάποιες ταξινομούνται ως τέτοιες και χωρίς να εξετάσουμε πολύ ενδελεχώς. Είδαμε κάποιες οργανώσεις που είχαν συσταθεί από κυβερνητικούς φορείς και ονομάζονταν μη μικρόν, όπως μια οργάνωση στην Κένια που ονομαζόταν κυβερνητική επιχείρηση για τους υδάτινους πόρους ή από κράτο μέλος που είχε συσταθεί από την κυβέρνηση υπό την τεχνική σκοπιά μπορεί και να είναι μη κάπα αλλά ε, δεν εμπίπτει στο πνεύμα του ότι πρέπει να είναι μη κάπα εφόσον από πίσω της είναι η κυβέρνηση. Και βεβαίω υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στο πώς ορίζονται και πώς αντιμετωπίζονται οι μη κάπα το οποίο έχει αντίκτυπο προς την λογοδοσία σε τρίτες χώρες. Γιατί σε κάποιες χώρε ταξινομούνται ως τέτοιες, σε άλλες όχι. Και σε τέτοια περίπτωση ίσως να έχουμε τελείως διαφορετικές απαιτήσει διαφάνειας ή υποβολής εκθέσεων. Τώρα προχωρώ στους κυριότερους αποδέκτες ενίσχυσης χορηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα νωρίτερα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια αξιόπιστη ανάλυση μέσω του συστήματος δημοσιονομικής διαφάνειας, του FTS. Από τις δεσμές 17, το 89% των χορηγιών δεν είχαν κανένα είδου οντότητα. Και στο 11% όπου διδόταν, δινόταν η οντότητα, υπήρχαν διάφορες παρατυπίες και διάφορα στοιχεία αρκετά παράξενα θα έλεγα. επαρκεί τέτοια κρούσματα ώστε να αρχίσει να σκέφτεται κανείς κατά πόσο μπορεί να βασίσει μια ανάλυση σε αυτά τα στοιχεία, σε τέτοιου είδους στοιχεία. Υπήρχε η αναδιανομή των ε, χορηγιών, το οποίο από ό,τι κατάλαβα ξεκίνησε και από ό,τι και νομίζουμε ότι του χρόνου θα γίνει συνολική εφαρμογή του αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο διανέμονται τα κονδύλια χορηγίας. Και καθότι δεν μπορούσαμε να έχουμε αξιόπιστο κατάλογο του top 30 των μη ομικρών από το FTS, λάβαμε ένα κατάλογο ε, που μας βοήθησε αρκετά από την γάμα budget, να πω ότι τα αποτελέσματα του καταλόγου αυτού είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα της προηγούμενης μελέτης, γιατί σε εκείνη τη μελέτη, εκείνη τη στιγμή μας είχαν ζητήσει να εξαιρέσουμε ερευνητικά Ινστιτούτα και πανεπιστήμια για τις δεσμεύσεις του 2017 που συμπεριελάμβαναν όμως τέτοιου είδους οντότητες. Εδώ Έχουμε τον κατάλογο του 17 με πρώτο ερευνητικό ίδρυμα αλλά και κάποιες πιο παραδοσιακά εννοούμενες ως μη είναι εκεί μεταξύ των πιο σημαντικών αποδεκτών. Αυτό είναι οι δεσμές του 15 και πάλι πολλά από τα ονόματα εδώ των οντοτήτων επαναλαμβάνονται στον κατάλογο του 17. Μας βεβαίωσε η ΓΔ Budget ότι θα μπορούσαμε να λάβουμε τα στοιχεία αυτά από ε, το FTS, αλλά δεν κατορθώσαμε να αναπαραγάγουμε τα αποτελέσματα που μας έδωσε η ΓΔ προϋπολογισμός. Και από αυτού πρέπει να πω ότι δεν μας απάντησαν τελικώς για την ανακολουθία αυτή. Τώρα στο Μητρό Διαφάνειας, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις έχουν αντίκτυπο στις μη όμικρον. Αυτή ήταν μια βασική ερώτηση. Στην προηγούμενη μελέτη είχαμε σημειώσει σειρά περιορισμών σχετικά με το Μητρό αυτό, που δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να το αναλύσει εύκολα λόγω της δομής και του είδους των πληροφοριών. Δεν ήταν δεσμευτικές, δεν ήταν εξακριβωμένες, πολλές δεν ήταν καθόλου αξιόπιστες και υπήρχαν και αποκλήσεις μεταξύ των όσων μπορούσαμε να ελέγξουμε και των όσων βλέπαμε ως καταχωρήσεις. Στην επικαιροποίηση η πληροφορία που είχαμε εμείς ήταν ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις τότε δεν είχαν συγκεκριμένο αντίκτυπο για τις ΜΚΟ, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον κάτι τέτοιο θα, καθιστούσε τα περιεχόμενα του Μητρώου πιο αξιόπιστα. και ίσως θα έπρεπε να αυξηθούν οι πόροι προς την γραμματεία που θα της επέτρεπε να προβαίνει σε περισσότερες εξακριβώσεις και να προβλέπονται ίσως και κάποιες κυρώσεις το οποίο βεβαίως και θα είχε αντίκτυπο σε μη καπαόμικρον αλλά όχι μόνο σε αυτές θα είχε αντίκτυπο σε οποιοδήποτε φορέα, οποιαδήποτε οντότητα καταχωρίζεται στο Μητρό Διαφάνειας. Και τέλος, από τις προηγούμενες συστάσεις είχαμε συστήσει ότι κάποιες από τις αποκλήσεις, μάλλον όλες, όλα τα σφάλματα ή όλες οι αποκλήσεις θα έπρεπε να αρθούν μέσω μιας κεντρικής τράπεζας δεδομένων. Η γάμα δέλτα budget μας είπε ότι το ABAC το σύστημα λογιστικής δεδουλευμένων είναι αυτή η κεντρική τράπεζα, αλλά στη σελίδα 8 έχουμε το μέγεθος 6 με μια καταχώρηση που καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο κεντρικό σύστημα, αλλά διάφορα συστήματα. Γιατί μας λέει ότι οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες για την αναδιανομή, ανακατανομή των ε, ε, κονδυλίων αυτών και παρακαλώ ελάτε σε επαφή με την ε, αρμόδια διεύθυνση κτλ. Το οποίο για μένα είναι σαφέστατη ένδειξη ύπαρξης πολλαπλών συστημάτων. Ενισχύει ακόμα αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχουν και οι εκταμιεύσεις που έχουν γίνει, οι συγκεκριμένες. και η αναδιανομή μεταξύ συμπράξεων ΜΚΟ ομικρών σχεδιάζεται από ό,τι κατάλαβα συνολικά ήδη από τις δεσμεύσεις του 18 και μετά και επομένως θα έπρεπε να είναι δυνατόν πλέον με τις νέες χορηγίες να δούμε πώς σχεδιάζεται αυτή η αναδιανομή. Είχαμε συμπεριλάβει μια μελέτη περίπτωσης στην περασμένη μας έκθεση για, τον, για την ερμηνεία των κριτηρίων εξαίρεσης. Και είχαμε πει ότι θα πρέπει να είναι πιο προδραστική η Κομισιόν παρακολουθώντας, επιτηρώντας τους πιο σημαντικούς αποδέκτες κονδυλίων. Υπό το φως πρόσφατου σκανδάλου βεβαίως υπήρξε ζωηρή δραστηριότητα σε αυτό αλλά δεν ξέρω αν αυτή η δραστηριότητα συνιστά συστηματική παρακολούθηση των πιο σημαντικών αποδεκτών. Απλώς ήταν προσπάθεια αντιμετώπισης ενός πολύ σοβαρού αλλά πολύ συγκεκριμένου κρούσματος το οποίο δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται μια γενικευμένη προσέγγιση διακυβέρνησης και η δημόσια ηχνηλασιμότητα και διαφάνεια σχετικά με την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν είδαμε κάποια κινητικότητα εδώ. Στην προηγούμενη μελέτη προσπαθούσαμε να παρακολουθήσουμε τα έργα όπως κατονομάζονταν στο σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας στις διάφορες ιστοσελίδες των δικαιούχων και σε μια τέτοια περίπτωση ήταν αδύνατο να βρούμε άλλη αναφορά στο όνομα υπό το οποίο είχε παραχωρηθεί το κονδύλι. Και ήταν δύσκολο ακόμα και όταν ξέραμε πού να ψάξουμε, τι ιστοσελίδες, τι ιστοτόπους, ήταν πολύ δύσκολο. Θα έλεγα σχεδόν αδύνατον να πούμε, μάλιστα, αυτή εδώ η δραστηριότητα που βλέπουμε τι σελίδες, τι τόπους χ, προέρχεται από την συγκεκριμένη δέσμευση ή κονδύλι που βλέπουμε στο FTS τάδε. Επ' αυτού κάναμε συστάσεις και κάναμε και συστάσεις για την επιφάνεια, την ε, ορατότητα των κονδυλίων αυτών, των χορηγίων αυτών. Η την έννοια τη είναι αδύνατο να έχει κανεί απόλυτη συμμόρφωση βέβαια, αλλά κάποιες φορές ε, σε ιστοσελίδα μετά από περίπλοκο και πολλαπλό κλικ πρέπει να πας πολύ βαθιά για να φτάσεις στα στοιχεία που χρειάζεσαι, αν είναι διαθέσιμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έλεγα ότι μια πιο συστηματική προσέγγιση χρειάζεται ώστε αυτού του είδους η ενημέρωση να είναι πολύ εμφανέστερη στις σελίδες των δικαιούχων και όχι μόνο για τις παρούσες χορηγίες, επιχορηγήσεις, όχι για τις τρέχουσες μόνο, αλλά και θα έπρεπε να υπάρχει ένα ιστορικό ώστε να φαίνεται, αν θέλετε, η ιστορική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δικαιούχους, στον κάθε δικαιούχο. Αυτά ήταν αυτά που ήθελα να σας πω που συνοψίζουν, νομίζω, την επικαιροποίηση στην προηγούμενη μελέτη που είχαμε υποβάλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η η κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα ε, περίμενα να πεις ότι φέρτε να πιούμε καναρακί εδώ πέρα όλοι, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Εντάξει, ωραία είναι η ενημέρωση και η επικαιροποίηση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε ε, και ε, που είχαμε επικρίνει και στο παρελθόν, ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και είναι πραγματικά έσχος και ντροπή. Εδώ πέρα στην Επιτροπή μας ασχολούμαστε με το να ακούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πόσο διαφανής είναι και πόσο καταπληκτική και θαυμάσια, ενώ ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι καθόλου ρόδινα όσο μας τα παρουσιάζουν. Το σύστημα χρηματοοικονομικής ε, διαφάνειας ε, είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκα στο προηγούμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή ε, και θα το επαναλάβω όμως, μπας και το χωνέψετε κάποια στιγμή. Ε, διαφάνεια δεν είναι να βλέπεις ποια κονδύλια έχουν δεσμευθεί ως ανάληψη υποχρεώσεων, αλλά και ποια έχουν εκταμιευθεί ως πληρωμές. Θέλω να ρωτήσω το συντάκτη της μελέτης, σας έδωσε κανένα λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν έχει συμβεί ακόμα αυτό και γιατί δεν είναι δημόσιο ποια χρήματα παίρνει ποιος και ποια γενική διεύθυνση ε, που χρηματοδοτεί με μονομένους δικαιούχους. Την ίδια ερώτηση θέλω να κάνω και προς προσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη σελίδα 18 βλέπουμε τους 30 μεγαλύτερους δικαιούχους. Και έχω μια ερώτηση. Στους πέντε πρώτους έχουμε δύο Γερμανούς, ένα Δανό, ε, δύο Δανούς και ένα Νορβηγό. Ε, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γεωγραφική ισορροπία έτσι κι αλλιώς. Αλλά Εκτός αυτού, γιατί παίρνουν τόσα λεφτά αυτοί, έχουν τα καλύτερα έργα ή ε, ε, κάτι που προκύπτει ιστορικά έπαιρναν τα περισσότερα λεφτά, πώς έχουν βγει τόσα εκατομμύρια εκεί. Και κάποια, ακόμα μια ερώτηση στο συντάκτη της μελέτης που μιλάει για τα δεοντολογικά. Με το σκάνδαλο Oxfam, το θυμάστε όλοι. Και στην προηγούμενη έκθεση ε, Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ έχει ε, ενισχύσει τα διοντολογικά και ηθικά κριτήρια. Αυτό στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Γιατί η μελέτη λέει ότι δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται αυτά τα πιο αυστηρά κριτήρια ή ε, πώς ελέγχεται η συμμόρφωση. Δεν θέλω να διαφωνήσω με τη βασική αρχή και σκέψη, αλλά αν καταλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επικεντρώνεται και βασίζεται πάρα πολύ σε δηλώσεις του δικαιούχου, εγώ δυσκολεύομαι να τα ε, πιστέψω. Κατά δήλωσή τους. Και ε, το αρμόδιο οργανό, γιατί δεν έλαβε την απόφαση να δημοσιεύονται αυτά τα στοιχεία. Είναι προς το δημόσιο συμφέρον, με άλλα λόγια. Αν δεν φτάνει ποτέ αυτή η πληροφόρηση στην κοινή γνώμη, τι σημαίνει. Ακόμα και όταν έχετε αποκλείσει, κάποιου, κάποιους από τη χρηματοδότηση, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν παίρνουν πια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και δεν δημοσιοποιείται τίποτα για τις τακτικές και τις πρακτικές τους, που μπορεί να είναι επιλήψιμες. Και πολλές φορές δεν τα δημοσιοποιούν ούτε οι ίδιες οι ΜΚΟ αυτά τα στοιχεία. Κρίμα, γιατί διαρριγνύουν τα ημάτια τους και απαιτούν πολλές ΜΚΟ ε, διαφάνεια απόλυτη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλες επιχειρήσεις πώς θα δώσουμε μεγαλύτερη προβολή και διαφάνεια στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φροντίσουμε να τηρούνται οι κείμενοι κανόνες. Αυτά και μακρηγόρησα. Δεν χρειάζεται να, προσθέσω ότι είμαι και απογοητευμένη ε, και σε απόγνωση από τη συγκεκριμένη μελέτη. Είναι καλή μελέτη γιατί είναι συγκεκριμένη και φωτίζει τις αδυναμίες ε, τη ε, κατάσταση. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα γιατί έχουμε και άλλο θέμα στην ημερήσια δέταξη. Okay, thank you. Uh, and this study very linked to the discussions we have. Ευχαριστώ πολύ. Οι μελέτες αυτές ε, τροφοδοτούν και τη συζήτηση που έχουμε κάνει εδώ. Ε, Ξεκινάμε κάτι θετικό. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η προσβασιμότητα και η ποιότητα των πληροφοριών για τι χρηματοδοτήσει αυτές έχει βελτιωθεί από το 2010 καθώς και από το 2016. Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να παρασχεί περισσότερες πληροφορίε για τους δικαιούχους χορηγιών επιχορηγήσεων και όπως εξήγησα ήδη έχουμε αλλάξει όλα τα συστήματα διαχείρισης ώστε να παρέχονται πλήρες πληροφορίες για τους δικαιούχους των κονδυλίων, όχι μόνο οι συντονιστές, αλλά και όλοι οι συνδικαιούχοι. Και σκοπεύουμε να κάνουμε το ίδιο και σε άλλους τομείς και ειδικότερα στις εξωτερικές δράσεις. Αυτό δείχνει πράγματι ότι έχει δεσμευτεί για διαρκή βελτίωση της διαχείρισης κομισιών όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ζήτημα το ζήτημα, όπως είπα προηγουμένως, είναι το πρόβλημα του ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το μόνο που ελέγχει το κεντρικό σύστημα της Κομισιόν είναι αν πρόκειται περί ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που ελέγχουμε. Μόνο αυτά μπορούμε να ελέγξουμε. Και αυτό και ελέγχουμε για όλους τους οργανισμούς που έχουν εγγραφεί στο λογιστικό σύστημα της Κομισιόν. Όπως υπόθηκε, ορισμένες φορές ε, υπάρχουν πανεπιστήμια και άλλες, κάποια άλλα. Όχι, ναι, πραγματικά κάποια πανεπιστήμια είναι μη και ιδιωτικά. Άλλα δεν είναι ιδιωτικά, είναι κρατικά. Πολύ λογικό λοιπόν που κάποια από αυτά συμμετέχουν, έχουν συμπεριληφθεί και κάποια άλλα όχι. Το βασικό ερώτημα είναι όμως, το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να επιληθεί αυτό το ζήτημα του ορισμού. Χρειαζόμαστε έναν ορισμό αποδεκτό από όλους. Και μετά μπορούμε να τον εφαρμόζουμε σε όλα τα διαχειριστικά συστήματα της Κομισιόν. Σημεία προβληματικά, διαφορετικά συστήματα ε, διαχείριση των επιχορηγήσεων είναι φυσιολογικό να έχουμε ένα σύστημα για την έρευνα, ένα σύστημα για τι εξωτερικέ δράσει. Αλλά μελετάμε αυτή τη στιγμή μια κοινή πόλη μεταξύ Κομισιών και των εξωτερικών ώστε να διευκολύνουμε τις ε, αιτήσει όλων των δικαιούχων όλων των αποδεκτών ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη διευκόλυνση των πληροφοριών μεταξύ αυτών και της Κομισιόν. Όσον αφορά την ε, προβολή, την ανακοίνωση, σύμφωνα με τη Μαλέτη, υπάρχει ανάγκη για πιο συστηματική προσέγγιση της ε, κοινοποίηση των δραστηριοτήτων που επιχορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεγαλύτερη προβολή. Πιστεύω ότι κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι σε όλες τις νομικές βάσεις που έχουμε εμείς προτείνει για το επόμενο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε εισάγει ένα άρθρο για την επικοινωνία και την προβολή που θα ισχύει όταν μια οντότητα λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια για την υλοποίηση ενός έργου. Αυτό έχει εισαχθεί σε όλες τις νομικές βάσεις για όλα τα προγράμματα του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όσον αφορά την δημοσιοποίηση των δικαιούχων ευρωπαϊκών κονδυλίων και την εισαγωγή των στοιχείων αυτών στι ιστοσελίδε. Ε, υπάρχει υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίε για τα έργα στην ιστοσελίδα. Αναφέρονται έργα που έχουν λάβει επιχορηγήσει από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούνται να εισάγουν όλες τις πληροφορίες, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να μπουν οι πληροφορίε στι γενικέ σελίδε του οργανισμού. Αυτό είναι σαφές ε, και στον δημοσιονομικό κανονισμό. Όσον αφορά αυτό που στις προηγούμενες συστάσεις, αυτό που έχουμε δει στις προηγούμενες συστάσεις, αυτό το 11% των δικαιούχων στο FTS ε, που έχουν ε, που έχουν κάποια ταξινόμηση. Ε, υπάρχει ένας κώδικας ε, σχετικός σε όλους τους δικαιούχους, αλλά υπάρχει και μια στήλη όπου μόνο αυτοί που έχουν δηλώσει ότι είναι ΜΚΟ έχουν τη σχετική ένδειξη δίπλα τους. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μόνο το 11%. Στις άλλες στήλες του ευθείας όμως μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες ε, των δικαιούχων και μπορούμε να δίνουμε και πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να εξηγούμε από πού προέρχονται αυτές τις πληροφορίες. Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών στο FTS. Μια άλλη ερώτηση αφορά τις εκταμιεύσεις του FTS. Το FTS ελέγχεται από την Δημοσιονομική Αρχή. Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να μπουν στο σύστημα του FTS θεσπίζονται στο άρθρο 38 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και όλες οι πληροφορίες που ζητά ο Δημοσιονομικός Κανονισμός δημοσιεύονται στο σύστημα ευθείας. Το μόνο που χρήζει ακόμα βελτίωση είναι η δεύτερη στρώση, το δεύτερο επίπεδο, οι δικαιούχοι δηλαδή της εξωτερικής δράσης, που αυτή τη στιγμή αναλύουμε. Η εκταμείευση δεν απαιτείται από τον κανονισμό, δεν ε, απαιτείται μόνο τα δεσμευμένα ποσά. Κύριε Άκερμαν, με δύο λόγια, πολύ σύντομα, γιατί έχουμε και άλλο θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Um, yes, I think, uh... Ε, πρόεδρε, Σας έκανε ερωτήσει η συγγήτρια. Oh, sorry. Already addressed to you. Σας έκανε ερωτήσει η συγγήτρια, απαντήστε. Um, ναι, κοιτάξτε, για τους πρώτους πέντε δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό, δεν είναι κάτι που εξετάσαμε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν έχω απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σμιτ. Τώρα επειδή δεν έχουμε χρόνο δυσκολεύομαι να ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Αλλά αυτό που είπε ο συντάκτη ε, δεν το ρώτησα εγώ. Δεν μου απαντήσει. Εγώ ρώτησα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σα έχει δώσει κανένα λόγο για ποιο. Καμιά δικαιολογία δηλαδή γιατί το σύστημα αυτό της δημοσιονομικής διαφάνειας δεν εφαρμόζεται ή της χρηματοδοτικής. Επίσης, σας ρώτησα για τις ηθικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις και τα κριτήρια μετά το κριτήριο της, και το σκάνδαλο μάλλον της Oxfam. Θα με ενδιαφέρει να μου απαντήσετε. Άμα γίνεται και αγαπρός, γραπτό, γραπτός δεν πειράζει αν δεν προλαβαίνετε τώρα. Και όταν κάνω ερωτήσεις μου αρέσει να μου απαντάνε. Για το θέμα της Oxfam θα ε, ζητούσα από τον εκπρόσωπο της ΓΔΕΚΟ ναι, ε, σα ευχαριστώ. Πράγματι, πράγματι εκπροσωπώ εδώ τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ε, Δημοσιονομικού Ελέγχου στην ΕΚΟ. Αυτό που κάναμε στην περίπτωση της Oxfam ήταν το εξής. Λάβαμε την ενημέρωση που όλοι έλαβαν το Φεβρουάριο και προχωρήσαμε σε μια παράλληλη στρατηγική, λέει ο Μελτής, αποστήλαμε έτοιμα ενημέρωσης από την Oxfam για το τι πραγματικά συνέβη το 2011 στην Αιτή και τους ζητήσαμε να περιγράψουν τα συστήματα που έχουν που είχαν πλέον το 18 δηλαδή για την πρόληψη και αποτροπή τέτοιων κρουσμάτων κατάχρησης. Αυτό κάναμε με την Oxfam. Παράλληλα όμως υποβάλαμε τις ίδιες ερωτήσεις για τα συστήματα σε όλους τους άνω των 200 εταίρους μας της ΓΔΕΚΟ. Στην απάντηση της Oxfam ήταν σαφές ότι χρειαζόμαστε περισσότερες διασφαλίσεις. Δηλαδή όχι μόνο επανεξέταση του συστήματος της, που χρησιμοποιούν δηλαδή εκείνοι, αλλά μια εξακρίβωση στο πεδίο ότι πράγματι το σύστημα λειτουργεί. Και γι' αυτό επισκεφθήκαμε μία από τις χώρες στις οποίες η Oxfam υλοποιούσε δράση της ε, γαμαδελταϊκός στο Λίβανο. Και ήρθαμε σε επαφή και με την έδρα της Oxfam στην Οξφόρδη. Προσπαθούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε τη λειτουργία των συστημάτων, τι ήταν αυτό που η Oxfam είχε εγγεγραμμένα στον κώδικα διοντολογίας της, κατά πόσον το σύστημά του λειτουργούσε επαρκώς, κατά πόσον ήταν εύκολα προσβάσιμο από τους δικαιούχους και το προσωπικό τους. Εξετάσαμε τη δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε περίπτωση κατάχρησης ε, ή εγκλήματος ή σεξουαλικής ε, εκμετάλλευσης και είχαμε, εν πάση περιπτώσει, ε, λογικά επαρκής διασφαλίσεις ότι είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν για να προλάβουν. Για τους υπόλοιπους 200 εταίρους ζητήσαμε την τις πληροφορίες αυτές και όταν δεν παρήχαν επαρκής, συνεχίσαμε να ζητούμε τις υπόλοιπες, λέει ο Μίλτης. Παράλληλα δεν προχωρήσαμε σε νέα επιχορήγηση προς την Oxfam. Έχουμε λοιπόν κάποια διδάγματα από αυτές τις εμπειρίες. Η συμβασιακή μας πολιτική στη εκο είναι σαφής για να είναι οποιοδήποτε φορέας εταίρος να την ξέρουμε τη διαδικασία. Thanks. Δεν χρειάζεται τώρα να τα παριθμίσετε όλα. Και τώρα θέλαμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παρακαλώ, ε, στείλτε ένα γράμμα τι κάνατε για την όξυπνα. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε εδώ το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστούμε για τη μελέτη και την παρουσίασή της και πάμε στο επόμενο θέμα. Ειδική έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάγκη λήψης μέτρων. Ο κύριος Πάρτς είναι το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου που θα μας παρουσιάσει τη μελέτη αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καταπολέμηση της ε, απάτης ε, κατά την εκτέλεση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καταλάβετε καλύτερα τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τα συμπεράσματα και τις συστάσεις πρέπει να καταλάβετε το πλαίσιο. Τι σημαίνει σωστή διαχείριση της, του κινδυνού απάτης σε στρατηγικό επίπεδο από τον οργανισμό που φέρει την ευθύνη ενώπιον του Κοινοβουλίου και των φορολογουμένων. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σωστή η διαχείριση της απάτης ε, σε τρία τμήματα του κύκλου πρόληψη και απόκριση και διαχείριση είναι σημαντική η πρόληψη, όπως επίσης και η απόκριση είναι απαραίτητη για αποτελεσματικές ε, αποτρεπτικές δράσεις. Ε, όσο λιγότερο τιμωρείται και ανοιχνεύεται η απάτη, τόσο περισσότεροι ε, την προτιμούν. Αυτό μας λένε εγκληματολόγοι. Αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, δεν υπάρχει αποτρεπτικό μέσο. Επίσης, πρέπει να καταλάβουμε το πλαίσιο και το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες όλο και περισσότερο ανησυχούν για τις απάτες ε, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής έρευνας. Αληθεύει ή όχι. Δεν ξέρουμε, ίσω να μην είναι καλά ενημερωμένοι οι πολίτε, δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό ήταν η αφετηρία για το ελεγκτικό συνέδριο. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε τον έλεγχο που εστιάζεται στο επίπεδο στρατηγικής διαχείρισης του πώς δηλαδή πραγματοποιείται αυτή η διαχείριση στρατηγική και πώς έχουν τα πράγματα σήμερα σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι είχατε μια μεγάλη μέρα σήμερα, αλλά ήθελα να σας τονίσω τέσσερα κομμάτια αυτής της έκθεσης. Έχουμε χρόνο. Α, ωραία. Τέσσερα ζητήματα είναι τα σημαντικά. Πρώτον, όσον αφορά το απάτη, όσον αφορά το αντικείμενο ε, τη φύση και τις αιτίες των απατών. Διότι οποιοδήποτε πρόβλημα με τη στρατηγική διαχείριση ξεκινά από την πληροφόρηση. Ποσοτική και ποιοτική. Αν δεν κατανοούμε το αντικείμενο, είναι αδύνατον να επιτύχουμε σωστά αποτελέσματα. Και τι ανακαλύψαμε κατά τον έλεγχο ότι η Κομισιόν δεν έχει επαρκείς πληροφορίες για την κλίμακα, τη φύση και τις αιτίες αυτό είναι το τρίγωνο που απαιτείται για την ε, καταπόλεμηση τη απάτη. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την ανείχνευση τη απάτη είναι ημιτελή. Προ το παρόν η Κομισιόν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία αξιολόγηση τη μη ε, σα απάτη. Βάσει αυτών των πληροφοριών που είναι ελλειπείς, πολλέ γενικέ διευθύνσει δηλώνουν ότι ο κίνδυνο απάτη είναι χαμηλό. Κατά την άψη του ελεγκτικού συνεδρίου, αυτό αποτελεί πλάνη. Πρώτα απ' όλα η Κομισιόν δεν συλλέγει επαρκείς πληροφορίες για το αντικείμενο, για το, πεδίο, για το εύρος της ε, και μετά λέει ότι είναι χαμηλό το επίπεδο. Αυτό είναι παράλογο. Όσον αφορά τις ε, ποιοτικές πληροφορίες που αφορούν ε, τα μοτίβα απάτης και τις αιτίες της απάτης, ούτε εδώ είναι καλύτερα τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμείς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κάποια τέτοια μοτίβα, κάποια συστήματα απάτης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά δεν πραγματοποιείται καμία ανάλυση που να μας βοηθήσει να καθορίσουμε το γιατί κάποιοι δικαιούχοι ευρωπαϊκών χρημάτων ε, επιλέγουν την απάτη. Σίγουρα δεν είναι όλοι απαταιώνε επαγγελματίε εγκληματίε. Για παράδειγμα, πολλέ μελέτε δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχει ε, κάποια σχέση αιτία αποτελέσματο μεταξύ τη απάτη και τη πολυπλοκότητα των κανόνων. Εξού και η πρώτη μα σύσταση προ την Επιτροπή. Το να δημιουργήσει ένα ε, ισχυρό σύστημα αναφορά των απατών που να παρέχει πληροφορίε για την κλίμακα, τη φύση και τι ε, ριζικέ αιτίε τη απάτη. Και θέλω να τονίσω, να επιστήσω την προσοχή σα, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ότι εδώ έχουμε και κάποιε διαφωνίε ε, με την Κομισιόν. Οπότε αναμένω τις ε, συζητήσεις ε, για να μπορέσουμε να σας εξηγήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τη λογική στην οποία βασίζεται αυτή η ιδέα ότι είναι σημαντικό να μελετάμε και τις μη ανιχνευθήσεις ε, περιπτώσεις απάτης και να έχουμε μια εικόνα για αυτές. Τώρα, όσον αφορά τα κίνητρα και το πνεύμα ηγεσία. Το ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίε ε, ε, στην Κομισιόν ε, δημιουργεί αμφισβήτηση όσον αφορά την πρακτική αξία των στρατηγικών σχέδιων, όπω τη στρατηγική καταπολέμηση τη απάτη, τη ΚΑΦΣΕ, που είναι η στρατηγική τη Κομισιόν. Αυτή, μάλιστα, η εταιρική στρατηγική δεν έχει επικαιροποιηθεί μετά το 2011. Οι στρατηγικέ καταπολέμησει τη απάτη στι γενικέ διευθύνσει που δαπανούν ευρωπαϊκά χρήματα επίση είναι αμφισβητήσιμε διότι χρησιμοποιούν κυρίως σλόγγαν για να περιγράψουν τους στόχους τους. Λένε ενίσχυση, ε, βελτίωση, ε, αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται συνήθως και συνήθως δεν δείχνουν ποιο είναι το σημείο αναφοράς, ποια είναι η αφετηρία και ποια είναι η τιμή στόχος, που θα ήταν προφανής πρακτική βάση των διεθνών προτύπων. που χρησιμοποιούνται ευρέω σε διάφορα οργανισμού ε, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η απάτη είναι ένα οριζόντιο ζήτημα και για την καταπολέμησή τη απαιτούνται συντονισμένε προσπάθειε πολλών μερών. Ταυτόχρονα το να καταπολεμήσει κανεί την απάτη δεν είναι. Η καταπολέμηση τη απάτη δεν αποτελεί βασική δραστηριότητα οποιοδήποτε τμήματο ή οργανισμού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια οντότητα κάποιο γενικό διευθυντή, ο οποίο να επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες αυτές ε, κατά πολέμηση της απάτης και με σαφείς ρόλους και ευθύνες στο προσωπικό, διότι αυτό θα βοηθήσει να αποφευθούν διπλές προσπάθειες ε, και να αξιολογηθούν ε, οι δράσεις του κάθε εμπλεκόμενου. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα η στρατηγική διαχείριση του κινδύνου απάτης και η πρόληψη της απάτης δεν αναφέρονται στο χαρτοφλέγιο κανενός επιτρόπου. Οι ρόλοι και οι ευθύνε των τμήματων της Κομισιόν που συμμετέχουν στις δράσεις καταπλέμησης της απάτης είναι κατακρεματισμένοι. Τα περισσότερα όργανα έχουν συμβουλευτικό ρόλο και η εταιρική επίβλεψη είναι ανεπαρκής. Αυτό μας οδήγησε στο να αντιληφθούμε ότι χρειάζονται περισσότερα κίνητρα και περισσότερο πνεύμα ηγεσία για να βελτιωθούν οι δραστηριότητε κατά πολέμηση τη απάτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν θα πρέπει να ξεκινά από ψηλά σε επίπεδο κολεγίου και να ε, να ορίσει έναν επίτροπο ω αρμόδιο για τη στρατηγική διαχείριση του κινδύνου ε, τη απάτη και την πρόληψη τη απάτη. Ε, το επόμενο ε, στοιχείο είναι ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα απόκριση. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σύστημα που να μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για πιθανού εγκληματίε ε, και να βοηθήσει σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείριση τη απάτη. Η αποτροπή λειτουργεί μόνο όταν εντοπίζονται οι απαταιώνε, διώκονται και τιμωρούνται επαρκώς με επαρκή κυρώσεις. Αυτό λέει ο νόμος. Αν δεν γίνονται διώξει, αν δεν τιμωρείται κανένας, τότε η αποτροπή είναι σαν να μην υπάρχει. Ο έλεγχος μας δείχνει ότι όλες οι έρευνες της Όλαφ Σπάνια αυτά καταλήγουν σε κάποια αποτελέσματα. Μόνο 17 διοικητικέ έρευνε τη Όλαφ κατέληξαν σε διώξει ετησίω. Και θέλω να σα το πω σαφέστατα. Το πρόβλημα δεν είναι το προσωπικό τη Όλαφ. Είναι υψηλά καταρτισμένο. Το πρόβλημα είναι το σύστημα. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα έρευνας και μετέπειτα δίωξης τα κράτη-μέλη απορρίπτουν πάνω από τις μισές υποθέσεις που προετοιμάζει η Όλαφ. Εδώ είναι και ο χρόνος. Παίζει σημαντικό ρόλο το σημαντικό σύστημα. Προβλέπει ότι η διοικητική έρευνα της Όλαφ πρέπει να ακολουθείται από ποινικές δύο έρευνες σε εθνικό επίπεδο. Μια τέτοια διαδικασία χρειάζεται χρόνο και καθιστά πολύ πιο αδύνατες τις περιπτώσεις δίωξης και πολύ πιο δύσκολες υπάρχει αυτή η εγγενής αδυναμία του συστήματος που δεν θα έρθει με τεχνικές βελτιώσεις στον κανονισμό της Όλαφ. Η εικόνα είναι το ίδιο άσχημη όσον αφορά την ε, ε, ε επιστροφή χρημάτων που έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί λόγο. Σε πολλέ περιπτώσει οι γενικέ διευθύνσει δεν βρίσκουν επαρκεί πληροφορίε για να ξεκινήσουν στι εκθέσει τη Όλαφ για να ξεκινήσουν τη σχετική διαδικασία. Ε, Επιστροφή των χρημάτων από το 2012 μέχρι το 2016 μόλις το 15% των συνολικού ποσού που ε, ανακάλυψε η Όλαφ πράγματι ανακτήθηκε. Έχουμε κάποιες αναλύσεις, αλλά δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε το διαιτητή εδώ και να πούμε ποιος κάνει τα πράγματα καλύτερα ή χειρότερα, αν είναι η Όλαφ ή οι γενικές διευθύνσεις. Από την άψη των φορολογουμένων δεν έχει σημασία ποιος δεν τα καταφέρνει πολύ καλά είτε είναι η Όλαφ είτε οι Γενικέ Διευθύνσει, διότι τα νούμερα δείχνουν ότι το σημερινό σύστημα δεν λειτουργεί καλά. Κατά την άποψή μα, και αυτή είναι η σύστασή μα όσον αφορά την Όλαφ, η Όλαφ ε, δεν μπορεί να λειτουργεί ω ε, ε, αστυνόμο που πραγματοποιεί έρευνε. Αυτή τη στιγμή μόνο υποβάλλει προτάσει σε άλλα όργανα προτάσει που δεν οδηγούν πάντα στα επιθυμητά αποτελέσματα, δηλαδή το να φέρουν του αποτελέσματα πρώτη δικαιοσύνη και να ε, ανακτήσουν τα χρήματα. Όπω είπαμε από την αρχή, η αποτροπή είναι το αποτέλεσμα ενό αποτελεσματικού συστήματο απόκριση. Αντί για αυτό, ο νομοθέτης θα πρέπει να δώσει στην Όλαφ ένα πιο στρατηγικό επιβλεπτικό ρόλο στην δράση καταπολέμηση τη απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πεπισμένοι στο ελεκτικό συνέδριο ότι χρειάζεται ένα οργανισμό που να σχεδιάζει την πολιτική αντιμετώπιση τη απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρακολουθεί την υλοποίηση αυτή τη πολιτική και να βλέπει πώ τα εθνικά συστήματα επιβολή του νόμου αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα τη περιπτώσει απάτη ευρωπαϊκών κονδυλίων που εμπίπτουν στι δικέ του αρμοδιότητες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοια συστήματα που να λειτουργούν σωστά. Στην έκθεσή μας επίσης δίνουμε και κάποια παραδείγματα για το πώς αυτός ο στρατηγικός ρόλος και η επίβλεψη θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Τι μορφή θα είχαν στα παραδείγματα του ΩΣΑ, αλλά αυτό μόνο ως έμπνευση για να δώσουμε κάποιες ιδέες. Πιθανότατα, αν και δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε εδώ, προσπαθούμε να περιγράψουμε πώς ο στρατηγικός ρόλος και η επίβλεψη ε, τι μορφή θα πρέπει να έχουν. Το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σίγουρα αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι αναμφίβολο. Ωστόσο, και στην έκθεσή μας ε, αναλύσαμε την νομοθεσία που έχει οθετηθεί και εντοπίσαμε κάποιους κινδύνους που μπορεί να εμποδίσουν ε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από όταν επιτύχει τους στόχους της. Ε, το πιο σοβαρό από αυτά τα θέματα είναι η ανείχνευση και η έρευνα ε, που εξαρτάται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών. Ο κανονισμός δεν έχει θεσπίσει κάποιο μηχανισμό που να δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να χωρούν πόρους απαραίτητους για την προενεργό ανείχνευση και τονίζω προενεργό ανείχνευση προδραστική ανείχνευση σοβαρών περιπτώσεων απάτης. Χρειάζεται να προλαμβάνουμε, να ανοιχνεύουμε τον των προτέρων την απάτη ω πιθανό κρυφό έγκλημα, λανθάνων έγκλημα υπάρχει σοβαρό, υπάρχει σοβαρός κινδύνος να μην φέρει καλά αποτελέσματα αυτός ο νέος θεσμός και το υπογραμμίζουμε στην εκτίση και θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προλαβαίνουν να εξετάσουν το θέμα και να αντιμετωπίσουν σωστά τους κινδύνους. Συμπερασματικά λοιπόν η πρόληψη, η ανείχνευση και η απόκριση στην απάτη δεν είναι επαρκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπερβολικά δύναμε. Η Κομισιόν δεν έχει σαφή εικόνα τη κλίμακα και των αιτιών τη απάτη. Το σύστημα επιβολή του νόμου δεν λειτουργεί σωστά και δεν ε, μα δίνουν τα χρήματα πίσω οι απαταιώνε. Δεν τα παίρνουμε πίσω από του απαταιώνε. Αυτή είναι μια ε, κατάσταση πολύ ανησυχητική και θέλουμε η Κομισιόν να αναλάβει δράση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι πράγματι έχει αναλυφθεί αυτή η δράση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι έτοιμος για να απαντήσω ερωτήσει. Ευχαριστώ κυρία Κινίτση. Συγγήτρια. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή τον κύριο Πάρτης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για την παρουσίαση, την εισήγηση που μας που σε έκανε για την ειδική αυτή έκθεση. Προφανώς εδώ μιλούμε όχι μόνο για υποχρέσεις που προβλέπουν οι συνθήκες, αλλά, αλλά κοινή ευθύνη για όλα τα κράτη-μέλη, γιατί όπως σωστά είπε ο πρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου, ανησυχούν οι πολίτες σχετικά με περιπτώσεις απάτης ή στις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πρέπει να δουλέψουμε ως προς την πρόληψη, πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψουμε ως προς μια ταχεία ανταπόκριση και αποτε... Ε, αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Είναι στην καρδιά δηλαδή της η ε, που πρέπει να αναλυθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι απατές. Τώρα, Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για να ενισχύσουμε την δυνατότητα της Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών να καταπολεμούν τις περιπτώσει απάτης. Αναφέρομαι στις διατάξεις ε, τι νομοθετικέ και όχι μόνο, στην ε, θέση ενισχύ του Early Warning Exclusion System, στην ε, μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού του 2018, στην υιοθέτηση της οδηγίας BIF και στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νομίζω ότι αυτές είναι διατάξεις, νομοθετικές προβλέψεις που θα μπορέσουν να δώσουν θετικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Όπως ακούσαμε βεβαίως ή στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, μας σημειώνονται κάποιες προβληματικές στοιχές του παράντος συστήματος που απαιτούν μια περαιτέρω εμβάθυνση και αναφέρομαι στις παρατηρήσεις του συνεδρίου σχετικά με την συλλογή και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων πλευράς της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τη ΟΛΑΦ για την αξιολόγηση κινδύνου στις διάφορες περιοχές δαπάνη. Επίσης αναφέρομαι στην σχετικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος έγκυρης προειδοποίησης και στις άλλες παρατήρησεις που ακούσαμε για την ελληματική παρακολούθηση την νομοθετική των συστάσεων όλα σε εθνικό επίπεδο οι οποίες πραγματικά θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε ε, αχίλιο πετέρνα της, ε, του συστήματος ε, αποτροπής απατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη γνωρίζουμε ότι δεν παρακολουθούν νομοθετικά σε άνω των 45% των περιπτώσεων που διαβιβάζει όλα και αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να μας ανησυχήσει. Η Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα στρατηγική κατά της απάτης που κανονικά θα πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτές τις ελλείψεις που σημειώνει το συνέδριο. Και στο πλαίσιο αυτό θα είναι χρήσιμο, πιστεύω, για όλου μα να έχουμε περαιτέρω πληροφορίε από την Κομισιόν για τον χρονοδιάγραμμα και το κυρίω περιεχόμενο του εγγράφου αυτού. Δηλαδή, αυτή η νέα στρατηγική κατά τη απάτη θα έχει επαρκεί χρηματοδοτικού και ανθρωπίνου πόρου. Για να έχει δηλαδή τη δυνατότητα που χρειάζεται και που σημειώνει ο Όλαφ για να αντιμετωπίζει τα κρούσματα απάτης η το των παρατηρήσεων του ελεκτικού συνεδρίου είναι απαραίτητο επίση να πούμε το εξή. Σχετικά με την περιορισμένη αποτελεσματικότητα του Early Warning System για τα κρούσματα χρηματοοικονομικής απάτης, από το 2016 ο δημοσιονομικό κανονισμό επιτρέπει όχι μόνο τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα, αλλά και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν την, την συγκεκριμένη τον φορέα ή επιχείρηση υπό την οδηγία PIF αρμόδιοι λοιπόν του συγκεκριμένου φορέα θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια, στην σύσταση νέου νομικού προσώπου και έτσι να παρακάψουν τον έλεγχο ή τις κυρώσεις. Αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός υπό την διοικητική και την προληπτική έννοια, αλλά στο ποινικό επίπεδο η νέα οδηγία, επικαιροποιημένη οδηγία ΠΙΦ δηλαδή, δεν συμπεριλαμβάνει πλέον συγκεκριμένη ρήτρα για την ευθύνη των επικεφαλής επιχειρήσεων. Σε σχέση με δράση ή δραστηριότητα που αναλαμβάνεται από υπάλληλο ή υφιστάμενο της επιχειρήσης εκείνης. Και επομένως αυτά θα μείνουν υπό τις εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας που όμως ε, όπως δείχνει πρόσφατη μελέτη υπό το Hercules 3 είναι τόσο αποκλίνουσες ώστε να δημιουργούν κενά ατιμορρησίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της υλοποίησης της οδηγίας ΠΥΦ. Ρωτώ λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο και την Κομισιόν η έλλειψη εναρμονισμένων και συγκεκριμένων διατάξεων σχετικά με τους επικεφαλείς επιχειρήσεων δεν είναι μια κρίσιμη έλλειψη, ένα κρίσιμο κενό για την πρόσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η έκθεση του συνεδρίου περιγράφει και κάποιες, μάλλον εκφράζει κάποιες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της μελλοντική ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Και επ' αυτού είχαμε όλοι μας ε, συζητήσει την πραγματικά περίπλοκη δομή που προβλέπεται για τον φορέα αυτό υπό τον κανονισμό σύστασης. Είναι απολύτως απαραίτητο για να ξεπεράσουμε τις ανησυχίες αυτές και τα ερωτηματικά, όχι μόνο να έχει η Ευρωπαϊκή Συγγελία επαρκή ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, αλλά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο να εγγυηθούμε δικαστικούς υπαλλήλους υψηλωτά της ακαιρεότητας και επαγγελματισμού. Αλλά έναντι των παρατηρήσεων που ακούσαμε από το ελεκτικό συνέδριο, θα πρέπει πέραν αυτών η Εβραϊκή Εισαγγελία να έχει άμεση και στενή συνεργασία με τον Όλαφ ο οποίο θα πρέπει να διατηρεί έναν στρατηγικό ρόλο ιδιαίτερα υψηλή σημασία. Ο Όλαφ παραμένει πολύ σημαντικό εταίρο συνεργάτη τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπορεί να διενεργεί επιπρόσθετε έρευνε. Υπό το άρθρο 21.3 του συστατικού κανονισμού της ακριβώς εισαγγελία. Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε επάρκειας προσωπικό ξαναλέω επαρκέ νομοθετικό πλάσιο, ώστε όλα αυτά να μπορεί να αντεπεξέλθει των δραστηριοτήτων αυτών, των καθηκόντων αυτών. Και μέσω της δραστηριότητός του και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορέσει στο μέλλον να καλύψει κάποια από αυτά τα κρίσιμα κενά που εντοπίζονται από το ελεγκτικό συνέδριο κάτι ακόμα να πω για την έλλειψη παρακολούθησης από πλευράς κρατών μελών για τις ε, συστάσεις ε, του Όλαφ και το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί μέσω της συμπερίληψης των πορισμάτων του Όλαφ σε περιπτώσεις και αστικού και ποινικού δικαίου. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια λύση ώστε να αυξήσει το επίπεδο αποτελεσματικής παρακολούθησης των κρατών μερών προς τις συστάσεις του Όλαφ. Η χρησιμοποίηση, για παράδειγμα, των στοιχείων που υποβάλλεται από τον Όλαφ ως αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσε να συμβοηθήσει τις εθνικές αρχές χωρίς να χρειάζεται να γίνονται και επικαλύψεις και να υπάρχει και αλληλοβοήθεια στο ανακριτικό και ερευνητικό έργο των αρχών. Σχετικά όμως με το αποδεικτό των στοιχείων αυτών που υποβάλλονται από τον Όλαφ θα πρέπει να υπάρχουν και επαρκείς ε, δικονομικές εγγυήσεις και στις ε, διοικητικές διαδικασίες και νομίζω ότι και, ο, και η Κομισιόν είναι απολύτως διατεθειμένη να δώσει αυτές τις ε, δικονομικές δικαστικές εγγύησεις. Τώρα, πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικότατο να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο για να προλαμβάνουμε την περι... τις περιπτώσεις απάτης, να λειτουργούμε ταχύτερα και να λειτουργούμε και προς την ανάκτηση των ποσών εκείνων, των κονδυλίων εκείνων, που στο τέλος λείπουν από τις στοχεύσεις που είχαν αρχικά στις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ όλους ε, για τη συνεισφορά τους εκ των προτέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Διερμηνία έχουμε μέχρι τις παρα 25 και μετά δυστυχώς τα αγγλικά τα υπόλοιπα. Ζητώ συγγνώμη κυρία Κινίτσι, προσπάθησα να ενθαρρύνω την Ιταλική καμπίνα να παραμείνει. Ε, αλλά δεν τα κατάφερα. Και τη γερμανική καμπίνα σταμάτησα να την ακούω. Κάποια στιγμή κόπηκε η διερμηνία, σταμάτησε στη μέση της πρότασης. Ωραία. Ε, ο συνάδελφος Τάραντ. Και 35 θα έχω τελειώσει, πρόεδρε, εντάξει. αλλά δυστυχώς μέχρι τότε έχω να πω πράγματα. Ε, γενικά σχόλια. Φαίνεται να είναι φινοουγγρικό το θέμα. Ένας εστονός ε, μέλος του ελεκτικού συνεδρίου κατηγορεί τον Φιλανδό πρόεδρο ε, της Όλαφ, διευθυντή. Εδώ και καιρό και μετά από καιρό έχουμε ευχάριστες ειδήσει από το ε, Λουξεμβούργο και τα διαβάζω αυτά στο πολίτικο. Από το ελεγκτικό συνέδριο ειδήσει δεν έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Και τώρα λέτε ε, ε, ότι είστε υπέρμαχοι των, ε, της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και κατηγορείτε τον Βίλε Ήταλ ότι δεν κάνει τίποτα για να πάρει τα λεφτά πίσω. Μα τα ξέρει, αλλά δεν μπορεί να επέμβει στις δικαστικές διαδικασίες των κρατών μελών. Το ελεγκτικό συνέδριο στο κείμενο χρησιμοποιεί όρους όπως μερικοί και συχνά, αλλά πολύ αόριστα, χωρίς να μας λέει συγκεκριμένα ποια είναι η έκταση και το μέγεθος του προβλήματος. Και αυτό θα πρέπει να μετρήσουμε. Όταν είσαι ελεκτικό συνέδριο, μετράς. Όπως γίνεται και στη φυσική. αυτό που κάνουν το δετερώνει, το νετρώνει. Αυτό που λέτε εσείς δεν είναι ευθύνη της Όλαφ, αλλά των κρατών μελών. Η ειδική έκθεση δεν αναγνωρίζει επαρκώ το στοιχείο αυτό και δεν επικρίνει καθόλου την αδράνεια των κρατών μελών. Έχουν ευθύνη όμως, την οποία δεν, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να υπερτονίσουμε. Και μιλώ στον κύριο Πάρτ τώρα, τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά και τον κύριο που κάθεται δίπλα σας, που είναι ο κύριο Κεν Μάρτι Βάχε. Εσείς τι κάνατε ακριβώς Ω μέλη ε, του ε, Συμβουλίου. Εσείς κύριε Πάρτσα έχετε διατελέσει πρωθυπουργός, εσείς κύριε Δίπλα έχετε διατελέσει υπουργός δικαιοσύνης. Τι έχετε κάνει για την Όλαφ ή μήπως τίποτα. το δεύτερο πιστεύω. Και ζητώ συγγνώμη και μάλιστα και λυπάμαι για την Εστονία που έχει τόσου κακούς εκπροσώπους στο Συμβούλιο. Και δεν φτάνει που τα κάνατε μουσκεμα, σας προήγαγα και σας έστειλαν στο Λουξεμβούργο. Σπουδαίο επίτευγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάω τώρα στα ειδικά σχόλια. Στην προηγούμενη ζωή σας παρεμποδίζατε οποιαδήποτε προσπάθεια κατά της διαφθοράς και της απάτης. Οποιαδήποτε ομοσπονδιακή εξέλιξη ως μέλος της ιστονικής κυβέρνησης. Και τώρα έρχεστε και κουνάτε και το δάχτυλο στον Όλαφ που επιτέλους και χάρη σε τούτο εδώ την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που εμείς συστήσαμε τον κύριο Βίλε Ήταλε, τον πρώην συνάδελφό σας στο Λουξεμβούργο, να γίνει Γενικός Διευθυντής στον Όλαφ. στο παρελθόν ε, κάνατε ό,τι μπορούσατε για να παρεμποδίσετε τον προκάτοχό του. Και τώρα έρχεστε και τον επικρίνετε. Και ειλικρινά ξέρω ότι η κυρία Κρέσλε θέλει να δώσει το λόγο σε άλλους για να πάμε σε άλλα σχόλια. Αλλά πριν τις 6.30 τουλάχιστον θα είχαμε κάνει κάποια, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Μην το παίρνετε προσωπικά, πολιτική είναι το θέμα και μόνο. Καλά, καμιά φορά μπορεί να είναι πικρή η επεξεργασία του παρελθόντος, αλλά σε αυτήν ε, ανήκει το να μην κατηγορούμε στο σημερινό Γενικό Διευθυντή για πράγματα του παρελθόντος και είναι συστημικά τα προβλήματα. Ούτε ο προηγούμενος φταίει. Και γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα ε, αυτή η έκθεση. Είναι η πρώτη έκθεση για την ε, λεγόμενη έκθεση PIF και πραγματικά μας ενδιαφέρει πολύ. Ο κύριος Νοβάκοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητά μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Ποιος θα πίστευε ότι στις 6.30 την Τρίτη το απόγευμα θα κάνουμε μία συζήτηση τόσο έντονη. Είμαι τυχερός που έμεινα μέχρι το τελευταίο σημείο και χαίρομαι που το επέλεξα αυτό. Σήμερα έχουμε μια σπάνια ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε για την Όλαφ δύο φορές μάλιστα. Πρώτον, συζητήσαμε την νομοθετική πρόταση της Κομισιόν. Την πρόταση που αφορά τις πιθανές σχέσεις ε, της Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, υπογραμμίζονται οι δυνατότητες της Όλαφ να εμβαθύνει τις ερευνές της εξέταζονται τα ενδεχόμενα επιπλέον ικανοτήτων, προσωπικού, μέσων, μηχανισμών, αναγνωρίζοντας ότι όλα προφανώς εξυπηρετεί το συμφέροντα των λαών μας ε, και ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να εκτελεί τι δραστηριότητε της. Όλοι ε, συμφωνούμε από αυτόν και με κάποια αντικειμενική κριτική. Και τώρα ξαφνικά έχουμε, το έχουμε γυρίσει από την άλλη. Επικρίνουμε την Όλαφ ότι δεν έχει αρκετά μέσα για τις έρευνες. Επικρίνουμε την Όλαφ ότι οι εθνικέ αρχές ε, δεν ακολουθούν τις συστάσεις τους. Έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιον ακούσω πια. Μέσα σε τέτοια σύγχυση αρχίζουμε να συζητάμε διάφορα. Μια από τις σημαντικότερες επικρίσεις στην έκθεση για την Όλαφ είναι ότι υπάρχουν αδυναμίες στη συνεργασία μεταξύ Όλαφ και εθνικών αρχών. Εδώ έχουμε δηλαδή δύο μέρη, την Όλαφ και τις εθνικές αρχές. Πρώτη ερώτηση, ποιες ε, ε, εθνικές αρχές ακριβώς, ποιος είναι ο ρόλος τους. Η εθνική νομοθεσία έχει να κάνει με την τήρηση των συστάσεων άλλη κριτική η δυνατότητα της Όλαφ να συγκεντρώνει επαρκή στοιχεία στο πλαίσιο ερευνών που να μπορούν να οδηγήσουν ε, συγκεκριμένους πιθανούς ε, εγκληματίες ενώπιον της δικαιοσύνης για να έχει τις ικανότητες η Όλαφ να εκτελεί αυτές τις ε, πράξεις καλύτερα Ποιο είναι το πρόβλημα αν ζητά περισσότερε θέσει εργασία ή αύξηση του προπολογισμού. Ε, σχετίζονται όλα αυτά. Εγώ είμαι αυτός που συχνά στο παρελθόν επέκρινα την Όλαφ. Όταν υπήρχαν αντικειμενικοί λόγοι. Τώρα όμω, ε, έχω την εντύπωση ότι κάποιε κάποιες από τις κριτικές ε, που εξαπολύουμε κατά τη ΟΛΑΦ δεν είναι δική τη ευθύνη, αλλά μια γενικότερη κατάσταση τη Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι ναι, η ΟΛΑΦ μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά αυτή τη στιγμή ε, και ειδικότερα τους τελευταίους ε, μήνες έχει δείξει η πολιτική ηγεσία τη βούληση, την επιθυμία να γίνει κάτι τέτοιο. Α εστιαστούμε λοιπόν στο πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι σχέσει μεταξύ Όλαφ και Εθνικών Αρχών, με ενδεχομένω κάποια ε, νέο ευρωπαϊκό νομοθέτημα ή βελτιώνοντα τη συνεργασία αυτή, ή δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο που θα βοηθήσει να. ενδυναμώσουμε όχι μόνο τις ευθύνες αλλά και τους μηχανισμούς που έχει στη διαθέσή της η Όλαφ για να παρεμβαίνει σε εθνικές υποθέσεις χωρίς απλά να τις επικρίνει για αποτελέσματα που εξαρτώνται καθαρά από τι εθνικέ αρχέ και που οι οποίε δεν υποχρεούνται να ακολουθούν τι ε, συστάσει, να βλέπουμε και τι δύο πλευρέ. Αυτό λέω. Οπότε εγώ έχω ελπίδα ότι αυτή η έκθεση σε τελική ανάλυση θα τροποποιηθεί επαρκώς ώστε να χαρακτηρίζεται από κάποια ισορροπία και πιθανότατα θα είναι και πιο αντικειμενική όσον αφορά τι δραστηριότητε τη Όλαφ, διότι όλοι συμφωνούμε εδώ ότι το ποσοστό σφάλματος μειώνεται και οι δραστηριότητε τη Όλαφ δείχνουν και οι εκθέσει τη Όλαφ δείχνουν ότι κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Για δεύτερη φορά σήμερα στην Επιτροπή μα, ο Γενικό Διευθυντή, ε, κύριος Έτελε, καλωσορίσατε με το επιτελείο σα. <laughs> Déjà Το έχουμε ξαναδεί το πρωί. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, όπω γνωρίζετε πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΟΒΕΡ έχουν μηδενική ανοχή για την απάτη και τη διαφθορά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την επιλογή του ελεγκτικού συνεδριού να ασχοληθεί με αυτό το σημαντικό θέμα. Στην έκθεσή του αναγνωρίζει τις προσπάθειες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα βήματα που αναλαμβάνει με την στρατηγική της πάταξης διαφθοράς και τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ελεκτικό συνέδριο και ο κύριος Πάρτς σήμερα φώτισαν κάποιους τομείς που χωρούν βελτίωση. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτά είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό τα περισσότερα και έχουν αντιμετωπιστεί ή αντιμετωπίζονται αυτό τον καιρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Όλαφ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Έχει εργαστεί σκληρά για την καταπολέμηση της απάτης τα τελευταία χρόνια, ε, μεταρρυθμίζοντας το ιστορικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου. Η Όλοφ διαδραματίζει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό και μοναδικό στη διερεύνηση και ανείχνευση πρώτα υπερεθνικών ε, περιπτώσεων απατών και διαφορά. Στα κράτη-μέλη, θυμίζω, είναι αρμόδια για την εκτέλεση των τριών τετάρτων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πρόληψη, ανείχνευση και διόρθωση ατασταλιών απατών και παρατυπιών. Πρόεδρε, πιστεύω ότι χρειάζεται σαφή δέσμευση από όλα τα κράτη-μέλη ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή αν θέλουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα ε, συμφωνούν με το ελεγκτικό συνέδριο ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για την καταπολέμηση της απάτης. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι περιπτώσεις απάτης ανοιχνεύονται και ερευνώνται ταχύτερα ε, σε όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια για να ενισχύσει το πλαίσιο καταπολέμησης της απάτης, όπως είναι η έγκριση της πρώτης στρατηγικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της απάτης, η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης ανείχνευσης και αποκλεισμού, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός. Η πρόταση ε, τροποποίησης του κανονισμού Όλαφ και η πρόσφατη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι άλλα στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή. Παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει στηθεί στα πόδια της και θα λειτουργεί μέχρι το 2020 και θα βελτιώσει σημαντικά τη συνέχεια που δίνεται σε περιπτώσεις απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα εθνικά δικαστήρια. Ο κανονισμός 883 που διέπει την όλα ενισχύεται και ε, ε, ε, διέπει καλύτερα του επιτόπιου ελέγχους στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, την πρόσβαση σε τραπεζικά ε, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και κυρίως στο παραδεκτό των ε, πιστήριων. Εδώ υπολογίζουμε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εγκριθούν αυτέ οι τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Όλαφ εργάζονται χέρι-χέρι για να βελτιωθεί και η ανάκτηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην πρόληψη της απάτης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τη στρατηγική της για τις εταιρείε και την αντιμετώπιση των απατών δίνει και ξέχοντα ρόλο στην Όλαφ σε όλη τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της απάτης. Για τις στατιστικές, για τις ατασταλίες παρατυπίες και την απάτη έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το σύστημα τα τελευταία χρόνια. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και εδώ σταματά η διερμηνία.